συζητήσουμε. Επιτρέψτε όμω να περάσω στη μέση ένταξη και δεν θέλω άλλο διαδικαστικό, παρακαλώ. Και τώρα. Είπαμε τη Δευτέρα. Έχετε την ημερήσια διάταξη, δεν αλλάζει τίποτα. Για τη Δευτέρα δεν υπάρχουν τροποποιήσεις. Τρίτη. Αρχίζουμε στις 9 το πρωί με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την διακοπή των ενέργειων μεταφορών στην Ευρώπη, 9 έως 11. Μετά 11 με 1 συζητούμε τα εξής θέματα. Δήλωση του Πρόεδρου Μπαρόσο σε σχέση με το νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010 και δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας στην IT. Δύο σημεία τα οποία είχαν προβλεφθεί από την αρχή στην ημερήσια διάταξη της ε, Τρίτης. Αύριο λοιπόν ψηφοφορίες δεν θα γίνουν, το μεσημέρι δεν θα γίνουν οι ψηφοφορίες. και ως προς τα υπόλοιπα η μερίσια διάταξη δεν αλλάζει. Προχωρώ στην Τετάρτη. Επίσης δεν γίνονται ψηφοφορίες Τετάρτη και αυτή είναι η μόνη αλλαγή σε σχέση με το ημερήσια διάταξη που έχετε μπροστά σας. Παραμένει η συνεδρίαση όλης της ημέρας ως έχει. Πέμπτη η σύνοδος δεν θα λάβει χώρα. Συνεδρίαση την Πέμπτη, σύνοδος μάλλον δεν θα γίνει. Ούτε ψηφοφορία δεν θα λάβει χώρα. Ούτε πρόκειται να γίνει συνεδρίαση που έχει προβλεφθεί για την απογευματινή συνεδρίαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η απόφαση της έσκεψη των Προέδρων ήταν παρόντες όλοι οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων, συμφώνησαν, ομόφωνα έλαβαν την απόφαση που σα ανακοίνωσα τώρα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη της σημερινή μας συνεδρίασης, η οποία τώρα προβλέπει τις μονόλεπτες παρεμβάσεις. Πριν να ξεκινήσουμε όμως, Θα ήθελα να κάνω την εξή ε, παρατήρηση. Δυνάμει το άρθρο 150, οι βουλευτές έχουν δικαίωμα σε παρεμβάσει ενό λεπτού. Από την εμπειρία μας όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν διπλάσια αιτήματα για τέτοιου είδους παρεμβάσεις από όσα θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε. Πολύ συχνά έχουν διατυπώσει τις διαμαρτυρίες τους ε, και την απογοήτευσή τους οι βουλευτές γιατί δεν είχαν το χρόνο που ήθελαν, δεν τους δόθηκε δηλαδή ευκαιρία να ομιλήσουν και για να αποφύγουμε περαιτέρω δυσαρέσεις και θα ήθελα πρότεινα το εξή για το μέλλον ως διαδικασία. Πρόκειται για τη διαδικασία που θα εφαρμόσουμε στις μονόλεπτες παρεμβάσεις. Δυνάμει του άρθρου 150 θα καταρτίζεται κατάλογος 30 ομιλητών με την, σεβόμενη την αρχή βέβαια της γεωγραφικής και πολιτικής ε, εκπροσώπησης και την προτεραιότητα κάθε φορά θα λαμβάνουν οι βουλευτές εκείνοι οι οποίοι στις δύο προηγούμενες ε, ε, συνόδους δεν είχαν, περίοδους συνόδου δεν είχαν λάβει τον λόγο για μονόλεπτη παρέμβαση. Όποιος δεν ε, λάβει αυτό το δικαίωμα της όλες παρεμβάσεως παρακαλείται είναι παρόν στην Ολομέλεια την ώρα που είναι η ώρα για αυτή τη συζήτηση και οι κανόνες οι οποίοι, σε τους οποίους σας εχθές θα σας αποσταλούν και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτές είναι ε, προτάσεις. Και ξεκινώ τώρα με τις μονόλεπτες παρεμβάσεις. Διαδικαστικό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου επιτρέπετε και παραλάβω το λόγο. Είναι πολύ περιορισμένο το χρονικό διάστημα που μας επιτρέπετε για να κοιτάξουμε τις εργασίες μας. Παρακαλώ λοιπόν να αναθεωρήσετε την απόφαση για ψηφοφορίες 5 και 6 Μαΐου. Οι Βρετανοί Ευρωβουλευτέ δεν θα είναι δυνατόν να είναι παρόντε την ημέρα των εθνικών μα εκλογών, των βουλευτικών μα εκλογών. Ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο θα απουσιάζει. Δεν μπορείτε να κάνετε ψηφοφορίε χωρί το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέσσερι του μηνό, παρακαλώ, να, να γίνουν οι ψηφοφορίε. Φέρτε λίγο πιο νωρί, παρακαλώ. Εάν ε, απορρίψω αυτό το αίτημα, αρνείστε και στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δυνατότητα να εκφράσει απόψει του. Να σα απαντήσω το εξή, λέει ο Πρόεδρο. Θα εξετάσω με την μέγιστη σοβαρότητα το αίτημά σα, κύριε συνάδελφε. Δύο είναι οι δυνατότητε που έχουμε, 5 και 6 Μαου και θα αποφασίσουμε το πώς θα χειριστούμε αυτή την υπόθεση των ψηφοφοριών. Είτε πέντε είτε έξι του μηγνώ και θα προσπαθήσουμε και να τις κατανείμουμε ενδεχομένω στις δύο ημέρες. Πρώτος μιλητής για τις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού είναι η κυρία Γιολάνα Χίπνερ. Ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μέλη του Σώματος θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ζήτημα των μεταλλαγμένων τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται προκειμένου να τροποποιήσει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου τα κράτη-μέλη να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία για να αποφασίσουν κατά πόσον θα καλλιεργήσουν ε, μεταλλαγμένα προϊόντα στο έδαφος τους. Προς το παρόν αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με βάση την νομοθεσία της ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν σύντομα θα υποβάλει πρόταση που θα επιτρέψει τα κράτη-μέλη να αποφασίζει τα, τα πόσον τα μεταλλαγμένα προϊόντα θα πρέπει να επιτραπούν. Πάντως, η απόφαση σχετικά με την εισαγωγή αυτών των μεταλλαγμένων προϊόντων είναι κάτι το οποίο ε, ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν ειδική επισήμανση και αυτές οι επισημάνσεις θα είναι πρέπει να είναι ιδιαίτερα σαφής και ξεκάθαρης προκειμένου ο καταναλωτής να γνωρίζει κατά πόσον τα προϊόντα τα οποία αγοράζει περιέχουν ή μη μεταλλαγμένα προϊόντα, μεταλλαγμένα τρόφιμα. Κύριος Μπάουντι. Μπάουντερ. Ντομινίκ Μπόντερ. Ο κύριος Ουγγουρένου. Πρόεδρε, να υπενθυμίσω στο σώμα ότι πριν από ένα χρόνο ε, έγιναν ε, κάποιες ε, παραβιάσεις στην Μολδαβία από κομμουνιστές και εδώ και ένα χρόνο η κυβέρνηση της χώρας, της χώρας αυτής έχει δείξει την ευρωπαϊκή της έφεση. Χρειάζεται λοιπόν η Μολδαβία την άμεση βοήθειά μα την κατάργηση των προξενικών θεωρήσεων και θα ήθελα να αναφέρω επίση και την περίπτωση του Έρναστ Βανταριάν, ενό δημοσιογράφου ο οποίος συνελήφθη και καταδικάστηκε για έσχατη προδοσία. Νομίζουμε ότι πρόκειται για μια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητάω από τους ε, επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μολδαβία να πράξουν τα απαραίτητα προκειμένου να απελευθερωθεί Λόγω λόγο Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ζαρμπόσκα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραμματέα, κύριε Επίτροπε, ήθελα να πω κάτι για ε, κάτι άλλο. Είχα προετοιμάσει κάτι άλλο να πω και τώρα το αφήνω στην άκρη. Ξέρουμε ότι έχουμε έκτακτα γεγονότα. Ε, λείπουν πολλοί συνάδελφοι, λείπουν πολλοί υπάλληλοι. Είχαν δυσκολευτεί πολύ κάποιοι άλλοι να φτάσουν μέχρι εδώ. Και αυτό θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτό το λεπτό που έχω στη διάθεσή μου ε, για να απευθυνθώ σε εσά κύριε Πρόεδρε και σε εσά κύριε γενική Γραμματεύ, κύριε Βέλε και να σας ευχαριστήσω πραγματικά φροντίσατε να μας εξασφαλίσετε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τις εργασίες μας. Από τις πρώτες ημέρες που ξέσπασε αυτό το πρόβλημα με την εναέρια κυκλοφορία, φρόντισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φτάσουμε όλοι στο Στρασβούργο, ε, να μας βοηθήσει όσο γίνεται και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εξ ονόματος συναδέλφων που είναι απόντες. Ο κύριος Μάρτιν για διαδικαστικό θέμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Και προηγουμένως προσπάθησα να τραβήξω την προσοχή σας όταν διαβάσατε τη νέα ε, ρύθμιση για τις μονόλεπτες τοποθετήσεις. Ακριβώς εσείς ως Πολωνός γνωρίζετε τι σημαίνει να υπάρχουν διάφορες κατηγορίες και τάξεις ανθρώπων και βουλευτών. Κοιτάτε λίγο και τα ορεινά έντρα να σας παρακαλώ. Επικοδομητικά τώρα, μπορείτε να μας εξηγήσετε ακριβώς τι είπατε προηγουμένω. Τι εννοείται δύο μήνε. Δύο μήνε στο Στρασβούργο ή και Βρυξέλλες μετράνε ε, πρώτη και ε, δεύτερη συνοδοση Στη συνέχεια. Τι θα κάνετε αν απουσιάζουν οι βουλευτέ που έχουν ζητήσει το μονόλεπτο για οποιοδήποτε λόγο. Θα δώσετε και κάτι στη ΔΙΑΗ. Και ένα τρίτο να ρωτήσω. Μπορείτε ήδη από σήμερα να διαβάσετε ποιοι είναι οι 30 ομιλητές που προβλέπονται για σήμερα στα πλαίσια αυτής της νέας ρύθμισης που την καλωσορίζω. Ε, dziękuję panu za Σας ευχαριστώ. Αυτοί οι κανόνες ε, θα εφαρμοστούν από την προσεχή συνεδρίαση στη συνέχιση των της Βρυξέλλες. Ο κύριος Φράιντρο έχει το έχει λόγο. Ο κύριος Λάξφριτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Από τις 15 ε, πρώτου το 2008 ε, ε, και είχε απαγορευτεί η θανατική ποινή μάλλον η σε κάποια θέματα μάλλον είχαν ξανάρχισε να θανατώνουν κάποια ζώα ε, ε, τα οποία όμως ε, προβλήματα αυτά συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων και, και τη μεταχείριση των ζώων θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ενδεχομένως στη ε, αλλά δεν συμφωνούν με αυτό. Και πρόεδρε τώρα έχουμε σε κάτι άλλο. Ε, θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας και πολύ επικοδομητικό να μας ενημερώνετε για συνεδριάσεις και συνόδους της Ολομέλειας νωρίτερα από ό,τι κάνατε ε, τώρα, γιατί η πρώτη μου πληροφόρηση ήρθε ε, την Κυριακή και δυσκολεύτηκα να φτάσω. Άμα σε ενημερώνετε νωρίτερα ότι θα, ε, ότι ξέρατε αυτό που θα συμβούν θα ήταν και περισσότεροι βουλευτές παρόντες. Αυτό προσπαθώ τώρα να σας εξηγήσω και το είπα και προηγουμένως. Ευχαριστώ. Θα σας απαντήσω αμέσως. τα σχόλια και τις παρατηρήσεις για τη σημερινή σύνοδο. Υπάρχει μια διαδικασία για το πώς λειτουργεί η Ολομέλεια και μόνο η σύνοδος ε, ολομελίας ή η διάσκεψη των Προεδρών είναι κυρίαρχη για να αποφασίσει εάν θα λάβει χώρα ή όχι, αν θα τροποποιηθεί. Γι' αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να συγκληθεί η συνεδρίαση αυτή στις 5 ε, το απόγευμα σήμερα ε, και να αποφασίσει το Κοινοβούλιο σε ολομέλεια. Ε, ε δεν προβλέπεται να μην συνεδριάζουμε καθόλου. Και ο κανόνας αυτός θα συνεχίσει να ισχύει για να ληφθεί μια απόφαση θα πρέπει να είναι απόφαση της ολομελίας ή να καταργηθεί ή να αλλάξει η προηγούμενη. να αλλαξει τώρα στις μονόλεπτες τοποθετήσεις και το λόγο έχει ο κύριος Κούτας. Când autorul noțiunii de produs intern brut uh, Simon Kuznets recunoștea că bunăstarea unei națiuni αναγνώρισε ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί ο πλούτος ενός κράτους από το ΑΕΠ του. Έχει όμως περάσει, χρειάστηκε όμως να περάσει ένας αιώνα ε, από την εποχή εκείνη μέχρι ότου βρεθούν οι κατάλληλοι μετρητές, οι κατάλληλοι δείκτες για να υπολογιστούν οι οικονομικές επιδόσεις των κρατών. Δεν είναι λοιπόν κατάλληλος δείκτης ε, το ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα γιατί δεν ε, ενσωματώνει την έννοια της ανάπτυξης και δεν καταγράφει και μορφές απασχόλησης όπως η εθελοντική εργασία. Προτείνεται λοιπόν ένα νέο σύστημα στατιστικής για την καλύτερη καταγραφή της ευημερία ε, των ε, πολιτών, καλύτερο υπολογισμό δηλαδή της ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι πια η εποχή κατάλληλη να καταμετρήσουμε την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη με ένα ενιαίο σύστημα για να καταγράψουμε και τα προβλήματα, τις κοινωνικές, τις κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπιλμπάου. Bilbao. Κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα ένα δικαστήριο όρισε ότι ε, το κλείσιμο της εφημερίδας Εγκουνκάρια στα βασκικά είναι αυθαίρετη πράξη άδικη και παράνομη και ορίζει η απόφαση του δικαστηρίου ότι και ούτε ο ποινικό κώδικας ούτε το Σύνταγμα της Ισπανίας επιτρέπουν να κλείσει εφημερίδα και βασίστηκε ε, στη ανόητη παραδοχή ότι να υπερασπίζεσαι τη βασική κουλτούρα σημαίνει ότι υποστηρίζει την ΕΤΑ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ανεξάρτητοι. Ούτε είχε ποτέ καμία σχέση χρηματοδότηση από και προ την ΕΤΑ. Ε, ήταν ε, μια διαδικασία που χόλαινε, ε, υπέστησαν βασανιστήρια και κακή μεταχείριση οι τη της εφημερίδας αυτής που ήταν σε κράτηση. Βλέπουμε δημαγωγία, διαχείριση της πληροφορίας, χειραγώγηση της κοινή γνώμης με συναισθηματικό τρόπο. Εμείς ε, είμαστε αντίθετοι με αυτή την αδικία και παρακαλώ να κλείσει με τρόπο δίκαιο αυτή η υπόθεση και να δικαιωθούν τα θύματα. Ευχαριστώ κύριο Στρεμόπουλος παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε τον ε, φεβρουάριο τον περασμένο παρουσιάσαμε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο την έκθεση ε, reuters trautmann της ευρωπαϊκής επιτροπής σχετικά με τις παγκόσμιες παράνομες αγορές ναρκωτικών από το 1998 και μετά. αυτή η έκθεση είναι μια πολύτιμη βάση δεδομένων και τα συμπεράσματά της επιβεβαιώνουν κάποιες αξιολογήσεις που υπήρχαν μέχρι τώρα για την μη αποτελεσματικότητα των πολιτικών περί ναρκωτικών στην ευρωπαϊκή ένωση αλλά και παγκόσμια. το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι τρέχουσες πολιτικές έχουν αποτύχει στον κύριο στόχο τους δηλαδή να μειωθεί η ζήτηση και προσφορά των παράνομων ουσιών ενώ αποτελούν ένα κρίσιμο παράγοντα αύξησης της βλάβης στους μεμονωμένους χρήστες το περιβάλλον τους την οικονομία και την κοινωνία. Ε, το 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα πακέτο συστάσεων όπως η έκθεση Κατάνια. Ζητούμε λοιπόν να ξαναδούμε το θέμα αυτό ε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ούτως ώστε να μην υπάρχει βλάβη um. Ευχαριστώ. Δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος, ο κύριος Τσενέτσκι. Ευχαριστώ. Ο λαός μου ε, θρηνεί, έζησε μια μεγάλη τραγωδία. Ο πρόεδρος της χώρας, ε, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, οι ε, ηγέτες από την πολιτιακή ηγεσία και τη στρατιωτική ηγεσία έχασαν τη ζωή τους. Εχθές εκειδεύτηκαν ο πρόεδρος της χώρας και η σύζυγός του. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκφραση αλληλεγγύης από πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης πραγματικά αποδείχθηκε τώρα στην πράξη. Για μας τους Πολωνούς ήταν υψή τη σημασία αυτό. Ο πρόεδρος της Αιχίας, της Σλοβακίας, της Γερμανία, της ρουμανία της Σλοβενία, και για να αναφέρω και λίγους μόνο ε, ήταν παρόντες στην κηδεία και ο Πρωθυπουργό της Εστονίας. Λυπάμαι προσωπικά που ο προεδρεύων του Συμβουλίου και ε, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κατάφερε να παραστούν. Αλλά ο πρωθυπουργός του Αζερβαϊτζάν και ο πρωθυπουργός της Γεωργίας παρευρέθηκαν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, παρευρισκομένους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερ Μάρτιν έχει το λόγο τώρα, αλλά δεν είναι εδώ. Απεχώρησε. Κύριος Μιόλτσας. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να κάνω κάποιε παρατηρήσει για τη Σερβία μέσα σε ένα λεπτό. Οι φιλοδοξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι τη ε, Σερβία ε, δεν έχουν ε, καμία βάση. Παραμένει παραμένει η προστασία, διατηρείται η προστασία την οποία έχει η Σερβία προσφέρει στους υπεύθυνους για τις γενοκτονίες από το στρατό της, ενώ ταυτόχρονα η Τουρκία η οποία βρίσκεται πολύ μακριά από την ένταξη κάνει κάποιες προσπάθειες για την συζήτηση θεμάτων όπως η αρμενική τραγωδία η αρμενική νοκτομηνία. Στην ε, Σερβία όμως βλέπουμε ότι ενώ έχουν διαιρεθεί σε πολυεθνοτικά κράτη και σε διαφορετικά κράτη διάφορες εθνοτικές ομάδες, ε, θεωρείται και είναι μια χώρα που αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σερβία ε, τμήμα της Ευρώπης δηλαδή, του πολιτισμού της και της παράδοσής της, αντίθετα από ότι η Τουρκία. Και ναι, δεν πρέπει να διαπράξουμε το σφάλμα που διαπράξαμε σχέση με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την προορία ένταξή τους, αλλά πρέπει να ενταχθεί κάποτε. Ο κ. παπα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η πρόσφατη, εξά... η πρόσφατη εξάρθρωση ενός σημαντικού πυρήνα της τρομοκρατίας στην ελλάδα έρχεται να υπενθυμίσει ότι η βία και η απειλή των δημοκρατικών θεσμών δεν γνωρίζουν σύνορα δεν κάνουν διακρίσεις. και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τρέχουσα η οικονομική κρίση και η απεσιοδοξία που αυτή γεννά στους πολίτες θρέφει επιθετικότητα παράγει βία. η βία καταδικάζεται όποια μορφή και αν έχει δεν διαφωνεί κανείς αυτό από όπου και αν προέρχεται. εκεί που επίσης όμως πρέπει να συμφωνήσουμε και να δώσουμε περισσότερη έμφαση είναι η σημασία της πρόληψης αντί της καταστολής. γι' αυτό πρέπει να ιεραρχούμε ακόμη πιο ψηλά ζητήματα που αναφέρονται στο swift στο pnr στην ενίσχυση της europol και της eurojust. σε κάθε περίπτωση είναι καθοριστικό να διορθώσουμε τις χρόνιες κοινωνικές παθογένειες που αναπαράγουν τη βία να χτυπήσουμε τη φτώχεια και την ανέχεια. δεν υπάρχουν περιθώρια αδράνειας. την τελευταία φορά που οι ηγέτες της ευρώπης δίλιασαν μπροστά στις κοινωνικές προκλήσεις των δύσκολων οικονομικά καιρών η ήπειρος βυθίστηκε στο σκοτάδι του μίσους και του ολοκληρωτισμού. Πρόεδρε, εξωτιμή θα ήθελα να επισημάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο τι πολύ ανησυχητικέ εξελίξει προ ε, τι τιμέ ε, των πρώτων υλών στο ε, που έχουμε πολύ σημαντική παραγωγή όπως και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες για τις θέσει εργασία των απασχολημένων στη βιομηχανία μα, γιατί έχουν ε, εκτοξευθεί στα ύψη οι τιμέ των πρώτων ελών και ιδιαίτερω σιδηρομεταλλεύματο. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιε προσπάθειε για να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε ε, ικανοποιητικέ τιμέ με μακροπρόθεσμε συμβάσει. Το ίδιο ισχύει και για το χάλιβα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με τις πρόσφατες αναδιαρθρώσεις στη Χαλιβουργία μας έχουμε περιορίσει σημαντικά το κόστος και ε, καταργήσει θέσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι από το Duisburg απέστειλαν και στην ε, καγκελάριο Μέρκελ και στον πρόεδρο Μπαρόσο μια έκκληση να σταθεί στο πλευρό τους και παρακαλώ να εισακουστεί. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Πατ Δεκόπ Κάλαχερ. Πρόεδρε. Καταστράφησαν, καταστράφησαν ε, πολλές από τις καλλιεργίες μας ε, λόγω της ε, ηφαιστειακής τέφρας που απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και μπορεί να ξαναρχίσουν οι ε, ναέριες μεταφορές αλλά ξέρουμε ότι είναι πολλοί οι επιβάτες οι οποίοι έχουν υποστεί σημαντικό κόστος ε, για τα δωμάτια των ξενοδοχείων που χρειάστηκε να πληρώσουν επιπλέον ή και για την παραμονή τους σε περιοχές ε, που δεν έχουν την οικία τους. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για θεομηνία και ότι έγινε σταλμένη από το Θεό η τιμωρία αυτή της ηφαιστειακής τέφρας. Παρακαλώ όμως να λογικευτούμε και να κοιτάξουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ε, ε, κληθεί τώρα να πληρώνουν ποσά τα οποία δεν έχουν πρόχειρα. Δεν είναι εύκολο να καλύψει κανεί αυτά τα έξοδα τα επιπλέον. Είναι επίγον να βρεθούν οι λύσει και επίση θα πρέπει, όπω ορίζει και σχετική οδηγία, να εφαρμόζονται οι υποθέσεις και τα επίπεδα ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ευχαριστώ κύριο Μορκάντη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα ήθελα στο αυτό το <laughs> σώμα να προτείνω να προβλημαριστούμε σχετικά ε, με, την επιρροή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις κοινότητες, στους ανθρώπους κλπ. Να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε μία ε, ιδέα ε, παγκόσμια και οικονομική ή να ε, εξετάσουμε, να επανέλθουμε μάλλον στην εξέταση των προβλημάτων ανθρώπων. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι μόνο έτσι θα δώσουμε μια αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Λαμβάνω υπόψη την οδηγία για τις υπηρεσίες του 2006, λεγόμενη Μπολκενστάιν δεν νομίζω ότι θα πρέπει να θυσιαστούν υπέρ μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του παγκόσμιου συστήματο ε, ο πολιτισμό ε, και η φιλοξενία που χαρακτηρίζει τι ε, τοπικέ κοινωνίε. Νομίζω ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει αποτελούν μια πραγματική δίνουν μάλλον το πραγματικό νόημα της, του πολιτισμού και της φιλοξενίας και θα πρέπει να τι προσπιστούμε. Ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. ευχαριστώ. Ως διάπειρος ευρωπαϊστής ε, δεν είναι εύκολο να ζεις αυτές τις μέρες. Θα ήθελα να σας παραπέμψω σήμερα στο πρόβλημα της Eurostat. Διαπιστώθηκε ότι η Eurostat ήξερε πολύ καλύτερα τι συνέβαινε στην Ελλάδα από ό,τι νομίζει η κοινή γνώμη. Ορισμένες εκθέσεις ήδη από το 2002 έχουν ε, συγκαλυφθεί εν μέρη για να βγει μεγάλη έκθεση το 2008 και είναι τελείως ασαφές πού πηγαίνουν οι εκθέσεις αυτές, τι συνέπειες έχουν, ποιες επιπτώσεις και ποιος φέρει την ευθύνη τώρα για την αδράνεια και την ολιγορία και ποιος είναι υπόλογος. Και τα τελευταία χρόνια είχαμε μια ε, ε, κατηγορία προς την Eurostat ε, σκανδαλοθυρική, αλλά κάποιος που ασχολείται σοβαρά με την Eurostat θα πρέπει να ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πώς θα δίνει σωστά στοιχεία ε, για να έχουμε πλέον μια επαναστατική δημοκρατία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ η κυρία Καρβάλιο. Obrigada, Presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον μιας φυσικής καταστροφής που έχει απρόβλεπτες ε, επιπτώσεις. Η επιστήμη μας επιτρέπει να υπολογίσουμε, μάλλον δεν μας επιτρέπει να υπολογίσουμε και να μετρήσουμε τα αποτελέσματα των ε, εκπομπών αυτών ε, της τέφρας για τα αεροσκάφη. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί με αυτά τα ε, με αυτήν την τέφρα. Οι υπουργοί συνεδριάζουν σήμερα προκειμένου να εξετάσουν τι θα γίνει με, το μέλλον των αεροπορικών μεταφορών. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την αρχή της προφύλαξης. Η οικονομία μας ε, δεν μπορεί να ε, επιβληθεί στην ασφάλεια των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν να προσπίσουμε την ασφάλεια των επιβατών με βάση κάποιες αποφάσεις ε, εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς και, του χρόνου, και άλλες χρονιές αντιμετωπίσαμε παρόμοιες ε, κρίσεις. Η πρώτη διακόπτη. Ε, λυπούμε, αλλά δεν έχετε πια άλλο χρόνο. Το λόγο τώρα θα λάβει ο κύριος Σέντσιου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στο τέλος του χρόνου πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή η τρίτη οδηγία για την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η χρηματοπιστωτική όμω κρίση ξέρουμε ότι επηρέασε και την ε, υπόθεση αυτή των ε, ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ε, προχωρεί λοιπόν η απελευθέρωση και ενισχύεται, βαθαίνει ακόμη περισσότερο η κρίση. Περιορίζονται οι ποιότητες των υπηρεσιών, περιορίζονται οι συναλλαγές και οι οι υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο πολίτης ακριβένουν τα τέλη και δεν παρέχονται επαρκή υπηρεσίε στι πιο απομακρυσμένε περιοχέ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να αποτρέψουμε την εμφάνιση ενό κοινωνικού ντάμπινγκ. Καλό δε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε μια ε, στην εισαγωγή ενός ορίου, μιας προθεσμίας μεταβατικής ε, δύο ετών για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρέντα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για τη δινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ερνέστ Μπαρντανιάν, ένας δημοσιογράφος ο οποίος ε, έχει φυλακιστεί στην υπερδυστερία από το εκεί καθεστώς. Ε, κατηγορείται μάλιστα για εσχάτη προδοσία, ε, για κατασκοπία. Βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και μόνο ε, οι αρχές του Τυράσπολ κάνουν μια χειρονομία προκειμένου να τον ε, να τον ε, στηρίξουν. Υπάρχει μια προσπάθεια να λυθεί η υπόθεση αυτή. Η τωρινή κυβέρνηση είναι υποτίθεται υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοευρωπαϊκή και καλό να απελευθερωθεί αυτός ο δημοσιογράφος ταχύτερο δυνατό και να προχωρήσουμε στο βαθμό που μπορούμε στη διευκόλυνση αυτών των ε, προβλημάτων. Ευχαριστώ κύριο Σικέρης και έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έπληξε περισσότερο τους πιο φτωχούς πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκριθεί στις περιστάσεις και στις ανάγκες. Γι' αυτό και το 2010 ε, ανακηρύχθηκε έτος πολέμηση της φτώχειας. 40 εκατομμύρια ε, πολίτες, σύμφωνα υπολογισμούς, είναι φτωχοί στην Ευρώπη και άλλα 40 εκατομμύρια απειλούνται ε, από τη φτώχεια. 20 εκατομμύρια είναι παιδιά. Είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μόνο ότι τους λείπει τροφή, φάρμακα, αλλά και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά τους λείπει και οποιαδήποτε προοπτική διεξόδου από το πρόβλημα αυτό. Για να αλλάξει αυτή η τραγική κατάσταση θα πρέπει να ποντάρουμε στην παιδεία πρώτα απ' όλα. Ιδιαίτερα ε, σε μικρές πόλεις και ε, στην Ήπεθρο χρειάζεται καταπολέμηση κατάσταση αυτής μέσω της παιδείας. Γι' αυτό χρειάζονται περισσότερες υποτροφίες και περισσότερα χρήματα εκεί. Ο κύριος Βόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αύριο θα εξετάσουμε το ζήτημα για ε, την αεροπορική κρίση, γιατί αυτό πλήττει όλους ε, τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, ιδιαίτερα τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει μια γενικότερη ύφεση. Κάποιες χώρες ε, έχουν κατορθώσει να βγουν από αυτή την ύφεση χάρη στις ε, κυβερνητικές πολιτικές ορισμένων κρατών. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία έχουμε στον Βασίλειο και τα οποία πρόκειται να ε, δημοσιευθούν τις προσεχείς μήνες. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ σημαντικό για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε περίπτωση κρίσης. Όλοι οι θεσμοί θα πρέπει να διασφαλίσουν πώς ε, θα μπορούν να υποστηριχθούν οι προϋπολογισμοί αλλά και οι πολίτες ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο κύριος Κούκαν είναι ο Κύριε Κουκάν. Δεν θα είναι εδώ μάλλον. Ο κύριος Φέιο παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει το ζήτημα των δημοσιονομικό που αφορά πολλά κράτη-μέλη. Αναφέρομαι σε αυτό το ζήτημα τη στιγμή που έχουν υποβληθεί οι προβλέψεις για μέσο μακροδοσμή περίοδο από ποικίλα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε σε ό,τι φορά την Πορτογαλία ότι το πρόβλημα αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζει κάποιους κινδύνους. Αυτό όμως ε, θα πρέπει να το πούμε λαμβάνοντα υπόψη την κατάσταση στην βρίσκονται τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Δεν μπορούμε να κοιτάζουμε μόνο το ζητήματα ανάπτυξης. Πάντως τα στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί από πολλά κράτη-μέλη δεν είναι διόλου ικανοποιητικά. Η ανταγωνιστικότητα, τα φορολογικά συστήματα, όλα αυτά συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Διαδικαστικό τώρα. Κύριο Ντόρτμουθ. Ε, ε, πάει καιρό που έχω ζητήσει τον ε, λόγο, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από τον συνάδελφο, ο οποίο μιλάει για παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να μα πει πώ εννοεί μια παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη ηφαιστειογενού τέφρα Ε, η Πρόεδρος, ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια των μονόλεπτων παρεμβάσεων δεν επιτρέπονται οι λεγόμενες παρεμβάσεις με, τη, με, τη, μπλε δελτίο, με την μπλε κάρτα. Εάν θέλετε διμερώς λύστε το, το θέμα, αλλά πάντως όχι μέσα, στη όχι μέσα στην Ολομέλεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα δεν έχουμε άλλο νομιλητή για τις μονόλεπτες παρεμβάσεις. Όσοι μπορούσαν να λάβουν το λόγο έχουν προκαταβολικά ε, ενημερωθεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην Ολομέλεια. Έτσι εξαντλήσαμε λοιπόν τον κατάλογο των εδώ παρόντων τουλάχιστον εγγεγραμμένων στον κατάλογο. Παρακαλώ, έχετε διαδικαστικό. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα σε ό,τι φορά την διαχείριση του λόγου να λαμβάνετε υπόψη την ισότητα ανδρών γυναικών. Ε, για πέντε φορές ε, συνεχώς δώσατε το λόγο σε άνδρα. Ευχαριστώ. Ως Προέδρος ε, της Επιτροπής Ψηλού Επιπέδου για την ε, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ασφαλώς θα, θα ε, φαντάζεστε και σωτητηρώ πάντοτε αυτό τον κανόνα. Απλώς μάλλον δεν ήταν παρούσες αρκετές γυναίκες για να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Αλλιώς το πράττουμε όποτε μπορούμε. Παίρνουμε στην ημερήσια διάταξη τώρα και πρώτη απ' όλα έχουμε την έκθεση του κυρίου Σάιον για την εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου. Το λόγο έχει ο εισηγητής πρώτος. Εξότιμε Πρόεδρε,